Κυρίε και κύριοι, θα θυμάστε ότι στι 6 Ιουλίου ε, κατά του κυρίου Κόρβιν Μίκ ε, επιβλήθηκαν κυρώσει για τι ε, ε απαράδεκτε παρατηρήσει του σε ό,τι αφορά Αφρικανού μετανάστε. Στι 7 Ιουνίου, ο κύριο Κόρβιν Μίκ υπέβαλε ένσταση κατά τη απόφαση αυτή και το Προεδρείο. Το Προεδρείο, συνεχίζει ο Προεδρό, εξέτασε την ένσταση και ομόφωνα επιβεβαίωσε την απόφασή μου. Με τις ε, κυρώσεις αυτές, λοιπόν, χάνει ο κ. Κορδημίκη για 10 ημέρες την ημερήσια αποζημίωση του και για 5 ημέρες αναστάλλεται η συμμετοχή του σε όλες τις κοινοβουλευτικές ε, δραστηριότητες πέρα από την ε, ψήφο του στην Ολομέλεια. Από τις 12 Σεπτεμβρίου, λοιπόν, θα ξεκινήσουν οι κυρώσει αυτές. Οι αρμόδιες Ιταλικές Αρχές με ενημέρωσαν για την εκλογή του κυρίου Άντζελο Τσόκα από τις 7 Ιουλίου. Ο κύριος Τσόκα θα αντικαταστήσει τον κυρία Τζον Λούκα Μπονάνο και καλώς ορίζω λοιπόν τον νέο συνάδελφο και να σα υπενθυμίσω ότι πλέον συγκαταλάγεται και μάλλον ε, ε, υποβάλλεται και πρέπει